Ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Θα ψηφίσουμε αύριο στο 12.30. Θα συνεχίσουμε την Ολομέλη αύριο, 25 Οκτωβρίου, 9 με 14, 15 με 22. Η ημερήσια διάταξη βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω να ευχαριστήσω τους διερμηνείς για την ευελιξία τους και διάθεσή τους. Πέρα στη συζήτηση.